Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του κανονισμού, ο πρόεδρος της διάσκεψης των ε, προέδρων με ενημέρωση για το εξή Δεν υπήρξαν κάποιες αντιρρήσεις για την σύσταση της Επιτροπής ε, ΕΚΟΝ για μία πράξη κατευσιοδότηση. Εάν ούτε μία ομάδα, ούτε τουλάχιστον 40 βουλευτές δεν εκφράσουν αντίρρηση εντός 24 ώρων ισχύει η σύσταση αυτή και ε, θα την βρείτε στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας. Οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές με ενημέρωσαν για αίτημα άρσης ασυλίας του κυρίου